Uh, Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Αλλά και από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες θα αργήσουν κάποιοι, γιατί έχουν άλλες συνεδριάσεις. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην σας ενόχλησε πολύ που περιμένατε. Ξεκινάμε τώρα, γιατί πήγε περίπου και 10. Θα τα πω αφού σας χαιρέτησα όλους στα αγγλικά, στη μητρική μου στα γερμανικά. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από πλευρά σας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εγκεκριμένη η μερίσια διάταξη. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Δεν βλέπω να θέλει κανείς κάτι να πει. Οπότε περνάμε στο σημείο 2. Η... Τα πρακτικά της συνεδρίασης τη 5 η Νοεμβρίου βρίσκονται στους φακέλους σα. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Και πάλι δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε προτείνω ότι ήθιστε τα πρακτικά να θεωρηθούν εγκεκριμένα εφόσον δεν προβληθούν αντιρρήσει ω το τέλος αυτή της συνεδρίασης. Περνάμε στο σημείο 3. Ανακοινώσει τη Προέδρου για τη διερμηνία. Έχουμε τις εξής γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, ουγγρικά, Λετωνικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και κροατικά. Και ήθελα ήδη να καλημερίσω τους διερμηνείς και να τους ευχαριστήσω που θα μας υποστηρίξουν σήμερα στη συνεδρίασή μα. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Σημείο 2, web streaming. Όπω θα γνωρίζετε, η συνάντηση αυτή μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Όπω τον διαγωγείο, θα έλεγα να έχετε καλή διαγωγή, αλλά τέλο πάντων καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και αποφάσει των συντονιστών 5 και 18 Νοεμβρίου 2019. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι ανακοινώσει των συντονιστών των δύο αυτών συνεδριάσεων 6 και 20 Νοεμβρίου έχουν μετα... Ε, αποσταλεί μέσω email στα μέλη της Επιτροπής ε, Κουλτ ε, για να τα εγκρίνεται και επισήμω μέχρι τις αντίστοιχες προθεσμίες 8 και 22 Νοεμβρίου. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις θεωρούνται εγκεκριμένες. Και μετά περνάμε στο σημείο 4. Η απαλλαγή του 2018, Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να το συνδυάσουμε με το επόμενο σημείο που αφορά το μεταφραστικό κέντρο και θα ήθελα να δούμε και τις δύο εκθέσεις, τις δύο γνωμοδοτήσεις μαζί και να τις συζητήσουμε από κοινού. Κυρίες και κύριοι, ε, για τα δύο σχέδια έκθεσης λοιπόν έχουμε μια διαδικασία απαλλαγής και για τους δύο τομείς, το γενικό προπολογισμό όπου έχουμε ευθύνη ως Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Παιδείας, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ ε, υπάρχουν πολλές δαπάνες που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας ή το Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Πολιτισμού και Παιδεία και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία επίπτουν επίση στο ίδιο πεδίο. Εδώ λοιπόν έχουμε ελέγξει τα στοιχεία του Erasmus Συν και έχουμε δει ότι ε, το πρόγραμμα αυτό έχει συμβάλει στην ευρωπαϊκή προσταθέμενη αξία με πολλού τρόπου. Βεβαίω, έχουμε μάθει από του υπευθύνου στα κράτη-μέλη ότι κάποιε φορέ οι εθνικέ συστάσει που πρέπει να ακολουθούν οι συμμετέχοντε δεν αντιστοιχούν στι απαιτήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση απολύτω. Γι' αυτό θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει τη συνέπεια των μέτρων εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη και να το παρακολουθεί το θέμα αυτό διότι δεν θέλουμε να υπάρχουν διαφορετικέ ε, εφαρμογέ ε, των ε, διαφόρων προδιαγραφών και προποθέσεων για το πρόγραμμα. Δυσκολεύουν τη συμμετοχή των φοιτητών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να διευκολύνουμε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα για να μπορέσει να υπάρξει και συνεργασία. Να μην γίνεται αυτή η περίπλοκη και μέσω της γραφειοκρατίας ε, πιο βεβαρημένη. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει εδώ επανειλημμένως και στην Επιτροπή μας. Και με αφορμή νέα προγράμματα πρέπει να είναι απλούστευμένη η διοικητική διαδικασία για την συμπλήρωση των εντύπων και για τη διαδικασία υπολογισμού και συμμετοχής. Πρέπει να γίνουν λοιπόν οι ανάλογες προσπάθειες με σχετικούς δείκτες για να δούμε κατά πόσο επιτυχάνονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Αυτό θα το δούμε και με αφορμή τα νέα προγράμματα που θα μας απασχολήσουν 2000, από το 2021, πώς μπορούμε να πετύχουμε βελτίωση. Ως προς τη διευκόλυνση για τους πολίτες, ε, για, τις, ε, για την υποστήριξη των φοιτητών, βλέπουμε δεν βλέπω εκπρόσωπο της Επιτροπής εδώ, αλλά έχουμε ίσως μια πρώτη φάση υλοποίησης που είναι πιο αργή. Θα πρέπει πάντως να εντοπίσουμε την ανάγκη αυτά τα προγράμματα να προχωρήσουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά αποφάσισε να πρικοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό με τα απαραίτητα μέσα. Ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χαιρετίζουμε την πρόβλεψη 11.000 θέσεων νέων ε, στο πλαίσιο του προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά στοιχεία για το πώς ελοποιήθηκε πρακτικά ε, το στοιχείο αυτό της πρακτικής εκδίπλωσης του προγράμματος. Θα έπρεπε να λάβουμε εδώ υπόψη πόσο στο μέλλον μπορούμε να ασχοληθούμε και με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις και να υπάρξει και η εθελοντική προσφορά, η εθελοντική συμμετοχή νέων, ώστε να ενισχυθεί το σώμα αλληλεγγύης. Είναι χρήσιμο για τους νέους που θέλουν εθελοντικά να ενισχύσουν το σώμα αλληλεγγύης. Για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe, υπάρχουν σοβαρά βήματα πρόοδου ε, σε σχέση με το διάστημα του 2007 31, 48% για το υποπρόγραμμα των μέσων και ενημέρωσης και 30% για τον πολιτισμό. Σε σχέση με το παρελθόν, λοιπόν, φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και τα αποτελέσματα αυτά δεν μα ικανοποιούν ακόμα πλήρω, αλλά ε, προφανώ υπάρχει ακόμα ανάγκη μεγαλύτερη χρηματοδότηση ή δυνατόν διπλασιασμό για την πυροδότηση του προγράμματο ε, Creative Europe. Όπω και στο παρελθόν, δυστυχώς έχουμε τα μισά από αυτά που ζητήσαμε και αυτό δημιουργεί απογοήτευση ε, και σε εμά ως υπευθύνου και στους συμμετέχοντες. Είναι λιγότερα από τα μισά αυτά που προσφέρονται ως κονδύλια. Οπότε το επαναλαμβάνω, θα πρέπει στου τριμερού διαλόγου και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να βρούμε τον ανάλογο προπολογισμό και για αυτά τα προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Πολιτισμό και την Παιδεία, Έχουμε διαπιστώσει ότι το εσωτερικό σύστημα ελέγχων πρέπει να βελτιωθεί με, τις ε, ανάλογες, με τους ανάλογους ελέγχους και στη δεύτερη φάση των ε, ελέγχων της δίκησης του προγράμματος Erasmus και Creative Europe. Ε, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες διόρθωσης με τα σχετικά μέτρα για να υλοποιείται καλύτερα το πρόγραμμα αυτό. Για τα ευρωπαϊκά σχολεία, το ελεκτικό συνέδριο εξέδωσε έκθεση τον Δεκέμβριο, ε, θα εκδώσει μάλλον έκθεση το Δεκέμβριο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τοποθετηθούμε για το θέμα αυτό αργότερα και να δούμε εάν υπάρχουν ανάγκε για αλλαγέ μετά την τοποθέτηση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Θέλω να σα ενημερώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λέγεται την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στι 4 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στι 21 Ιανουαρίου. Θα φροντίσουμε τον τω να οργανώσουμε και τι ανάλογε συναντήσει και οδών ηγητών για να συζητήσουμε όσα χρειάζεται. και να είναι σχετικά απλωστημένη η διαδικασία. Τώρα για το κέντρο μετάφρασης, ε, επειδή και αυτό περιλαμβάνεται στη δικασία απελάγης. είναι υπεύθυνο για την πολυγλωσία το κέντρο αυτό και ο τρόπος που λειτουργεί αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, όπως έχουμε διαπιστώσει από την προηγούμενη διαδικασία, αποφασίσαμε να δώσουμε την απαλλαγή Αν και κάποια στοιχεία για κάποιες γλώσσες έφτασαν αργότερα από άλλα, είχε ήδη εκπνεύσει το πρόγραμμα Εράσμους μέχρι να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σχετικές γλώσσες, οπότε αυτό δεν αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης. Πάντως πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε και με αυτόν τον τρόπο την ε, πολυγλωσία. Ε, είναι θετική η αποτίμηση του κέντρου μετάφρασης με 4,4 εκατομμύρια από το 2019 και πλέον το κέντρο, το κέντρο δείχνει ότι έχει ε, προσωπικό με υψηλά προσόντα, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω στη διοίκηση και το επίπεδο των μάνατζερ και θα πρέπει να προκοδοτηθεί με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της ψηφιοποίησης για τα προγράμματα αναγνώρισης της γλώσσας, για παράδειγμα, και το πρόγραμμα Ορολογία για την Ευρώπη, Terminology for Europe. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηριχθεί ε, για να ολοκληρώσει τα σχετικά προγράμματα που μέχρι το 2018 δεν είχαν περατωθεί. Σε ευρωπαϊκό λοιπόν επίπεδο πρέπει να αναζητήσουμε τους αναλογούς μηχανισμούς για να υποστηρίξουμε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης. Έχουμε λοιπόν εδώ χρόνο για ένα γύρο ερωταπαντήσεων και θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές και μετά στους υπόλοιπους ε, βουλευτές της Επιτροπής που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν. Παρακαλώ, αν θέλετε το λόγο, να το δηλώσετε για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε εδώ τον κατάλογο αγορητών. Ξεκινώ με τους σκιώδεις εισηγητές, η κυρία Φεγά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τη δουλειά σας ε, την πλήρη. Είναι δύσκολο βέβαια όταν κάποιο είναι νέος ε, βουλευτής να πάρει θέση για τον προπολογισμό του 2018. Σημείωσα πάντω ε, τις απόψεις ε, οι οποίες ε, είναι σχολαστικές ε, και πλήρεις. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πολυγλωσία για το κέντρο μετάφραση τη σχετική γνωμοδότηση είναι πολύ καλό το φέρετε, διότι αυτό φέρνει τη δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη και είναι πιο αποτελεσματική. Σε ό,τι αφορά ε, την προπολογισμό τη Κομισιόν, είναι η κλασική ε, διάρθρωση με το τσόμα αλληλεγγύης, το Erasmus Plus κτλ. Ε, εγώ θα ήθελα να προτείνω να αναφέρουμε για το 2018 και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς που χρηματοδοτήθηκε ε, ακριβώς για το... Ε, με ένα ποσό 8 ευρώ, δόθηκε δηλαδή ειδική χρηματοδότηση, πέρα από τη μελλοντική γνωμοδότηση πρωτοβουλία τη Επιτροπή μα, καλό θα ήταν να, το πούμε αυτό στη γνωμοδότησή μα ε, που θα στείλουμε στην Επιτροπή Κοντ. Είναι ένα σημείο που ήθελα να αναφέρω. Επίσης θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποιες αναφορές ε, στην ισότητα, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο κείμενο, διότι κάποια προγράμματα έχουν ε, αρκετά ενθαρρυντικά ποσοστά βεβαίω συμμετοχή των γυναικών, αλλά παραμένουν μακριά από την ε, ισότητα. Θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε και βεβαίω αναμένουμε την μονησία να συζητήσουμε στο μέλλον τη νομοδότησή σα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Λέκριος Λαμπάκοφ. Θα ήθελα να αναφερθώ ταυτόχρονα και στους δύο φακέλους. Είμαι σκιώδης συγητής και για, τα, για τους δύο. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι εγώ είμαι κατά αυτής της ψήφου πριν το ελεγκτικό συνέδριο εκδώσει τις εκθέσεις του. Ε, είναι αρκετά ατελής, δεν είναι πλήρης ε, η ε, πλήρη τα κείμενα αυτά σα διότι δεν έχουμε ακριβώς το πόρισμα του Ελληνικού Συνεδρίου. Ε, Βεβαίω εδώ δίνεται έμφαση στο Erasmus Plus ε, πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε η γραφειοκρατία όμως είναι εξαιρετικά προβληματικό αυτό ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού και του και της εκπαίδευσης χαίρομαι που γίνεται αναφορά στην δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολυγλωσία. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε μόνο τη γλώσσα των μεγάλων χωρών. Όλα τα κράτη-μέλη είναι ίσα και αυτό ισχύει και για τις γλώσσες. Εάν λοιπόν προωθήσουμε τα γαλλικά πρέπει να προωθήσουμε και τα λετονικά, τα βουλγάρικα. Διαπιστώνω όμως ότι υπάρχει διαφορά ε, στο κέντρο μετάφρασης. Ο στόχος ε, της καταπολέμησης της απάτης ήταν στο 66% έχουμε ξεπεράσει τη σχετική ποσόστοση για την κατάρτιση των υπαλλήλων αυτό μου φαίνεται πραγματικά περίεργο ανησυχώ επίσης ε, για τα χαμηλά αποτελέσματα ε, του Creative Europe δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά είναι σκανδαλώδες αυτή η εδαφική κατανομή τον project ε, είναι προβληματική. Ε, επίσης, ε, αν δούμε και τους δικαιούχους, τα στατιστικά στοιχεία δεν θα τα δούμε ποτέ και για το πρόγραμμα Media. Μόνο κάποιες, κάποιες εθνικές βιομηχανίες κινηματογράφου θα έχουν υποφεληθεί αυτών των προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Media. Μόνο σε κάποιες χώρες Λοιπόν, δεν είναι ικανοποιητικέ αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Πολύ σύντομα για το ελεκτικό συνέδριο. Η έκθεση για τα ευρωπαϊκά σχολεία αναμένεται. Τις υπόλοιπες τις έχουμε. Τον Γενάρη θα αποφασίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μέχρι το Δεκέμβριο να δημοσιευτεί η έκθεση αυτή. Σας βεβαιώ όμως ότι θα λάβετε τις ανάλογες πληροφορίες αυτό το χρόνο για την Επιτροπή θα, τοποθε... θα μας πει ο πρόσωπός της έτσι κι τη δική του στη Σκοπιά. Κάτι έγινε με την αγγλική μετάφραση, οπότε να τα πω αγγλικά. Α, τώρα δουλεύει. Να τα ξαναπώ. <laughs> <laughs> Ξεκίνησε ήδη το Brexit. Έλεγα απλώ στον συνάδελφο Σλάμπακοφ ότι η μόνη εκθέση που μα λείπει από το ελληνικό συνέδριο είναι αυτή που αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία. Το Δεκέμβριο θα τα λάβουμε. Οπότε το Γενάρη αποφασίζουμε να μην αναλόγω για να έχουμε και τα στοιχεία. Πρέπει να προσέξουμε να κανονίσουμε έτσι την προθεσμία για την υποβολή των απολογιών, ώστε να, μπορεί, έχετε χρόνο να δείτε και τις, λεπτομέρειε λεπτομέρειες του προγράμματος. Και θα μπορεί να μας πει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζομαι, να μας δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το θέμα. Και τώρα Θέλω να δώσω το λόγο στους συναδέλφους από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ή όποιον εκπροσωπεί τους και εισηγητές που δεν είναι παρόντες. Όποιον θέλει κάτι να πει. Hello. I would like to pick up on the... Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που έδωσε ο κύριος Λάμπακοφ για τα ποσοστά επιτυχίας 31% ε, για το CALT και 38% στα πλαίσια του Media για το Creative Europe ε, σε έναν άλλον φάκελο ε, μου εξήγησαν ότι το ποσοστό επιτυχίας δεν σημαίνει ότι το project ολοκληρώθηκε και ότι πήγε καλά ή όχι είναι πόσα, πόσες επιδοτήσεις, πόσες υποτροφίες δόθηκαν και πόσες αιτήσει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο. Ίσως για το θέμα των ποσοστών ε, επιδόσεων. Ε, γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Δεν μιλάμε για την επιτυχία του προγράμματος, μιλάμε για τις επιδόσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα. Δηλαδή, πόσοι από αυτού που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τελικά υποστηρίχθηκαν, έλαβαν υποστήριξη. Δηλαδή, εγώ ως ε, υπεύθυνος για το πρόγραμμα, από αυτούς που αναπτύσσουν το πρόγραμμα, κατά πόσον έχω κάποιο ποσοστό επιτυχίας, πιθανότητες να προχωρήσω για το Εράσμους. Εκεί μιλάμε για ποσοστά επιτυχίας κάτω του 20%, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα θεωρητικά, δηλαδή υποστηρίζουμε πολύ περισσότερα από πω ότι ε, στην πραγματικότητα επιδόσεις έχουν οι συμμετέχοντες. Θέλουμε δηλαδή να πούμε ότι ε, είναι λίγο παραπλανητικός ο όρος, διότι ε, έχουμε πάντοτε πολλά νέα μέλη που δεν τα γνωρίζουν, ενώ με ποσοστά επιτυχία στο κατά πόσο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε περισσότερους από ό,τι τελικά υποστηρίχθηκαν. Ο όρος λοιπόν ε, επιτυχιών έχει να κάνει με τις πιθανότητες ε, συμμετοχής στο πρόγραμμα ποιοι μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα. So in fact, this is actually a really good... Αλλά είναι πολύ καλός ε, ο αριθμός. Δείχνει πόσο επιτυχημένα είναι τα προγράμματα, πόσο ε, ε, πολύ συμμετέχει ο κόσμος. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Εάν όχι, να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την γνωμοδότηση. Ε, είναι πολύ ικανοποιημένη η Κομισιόν, όπως και εσείς, για τα αποτελέσματα των ελέγχων του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά το Erasmus Plus ε, και το ε, Σώμα Αλληλεγγύης. Ε, η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εδώ και πολλά χρόνια το ποσοστό σφάλματος βρίσκεται κάτω από το, από το κατόφλευτο του 2%. Επίσης, είναι ικανοποιημένη η Κομισιόν από τα αποτελέσματα της ε, ε, του ελέγχου απόδοσης, ε, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι ε, πολλαπλώς προκύπτει προστιθέμενη αξία. Το ελεγκτικό συνέδριο, όπως και εσείς αναφέρετε στην γνωμοδότησή σας, ζητάει καλύτερη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κατάρτισης και εκπαίδευσης. Άλλωστε, η Κομισιόν προετοιμάζεται για την νέα γενιά αυτού του προγράμματος. Επίσης, όσον αφορά αφορά τους ε, κανόνες ε, που δεν είναι ομοιογενώς εφαρμοζόμενοι στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ταυτοποιηθούν ε, με καλύτερο τρόπο όσοι έχουν ειδικέ ανάγκες και που προέρχονται από ε, περιβάλλοντα πιο ε, ευάλωτα ή μειονεκτούντα. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ε, ξεχωριστός υπολογισμός αυτών των ανθρώπων όσον αφορά τώρα την, τη νεα γενναια γενεά προγραμμάτων 2021-2025. Η Κομισιόν προτίθεται να ε, έχει μια, έναν νέο ορισμό ε, κριτηρίων που θα είναι πιο συγκεκριμένοι και που θα οδηγούν ε, σε μεγαλύτερη συνεκτικότητα του προγράμματος έρευνους επί τόπου όσον αφορά την ΕΚΑΕΑ. Είναι ικανοποιημένη η Κομισιόν για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται αυτή η υπηρεσία. Έχουμε ένα νέο διοικητή της υπηρεσίας αυτής και επομένως ένα νέο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα έχει στόχο την βελτίωση των, ε, του, του εσωτερικού, της εσωτερικής μεθοδολογίας εργασίας καθώς επίσης και την δυνατότητα να προσαρμοστεί ε, σε προγράμματα με μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο μέλλον. Βεβαίως θα υπάρξει και μια εσωτερι... ένας εσωτερικός οικονομικός έλεγχος, έλεγχος παρακολούθησης από τις εσωτερικές υπηρεσίες ε, της Κομισιόν. Ε, ε, πέρα από αυτό, ε, στις διοικητικές συνεδριάσεις της υπηρεσίας θα υπάρξει και εξωτερικός παρατηρητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω Τη σχετική γνωμοδότηση θα την ξαναδούμε το Γενάρη ε, και θα δούμε τις σχετικές απόψεις γιατί ε, θα έχουμε κενά εάν το κάνουμε από τώρα. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Τεχνολογικό Ινστιτούτο για τα θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας. Και τώρα να περιμένουμε την κυρία Χόφμαν στο Προεδρείο. Frau schön, dass Sie da sind. Ευχαριστούμε κυρία Χόφμαν που ήρθατε σήμερα. Ε, Όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας, μαζί με την Επιτροπή ΤΡΕ, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το σχετικό νομοθετικό πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη παρουσίασε ένα πακέτο για την ε, στρατηγική ατζέντα της καινοτομίας τον Ιούνιο για το διάστημα 2021-2027. Οι δύο συνεισηγητές μας, Έλερ και Μπάντινγκ, από το ΕΛΚ και την ΡΙΝΙΟΥ, ετοιμάζουν τα σχέδια γνωμοδότησή του και θα τα παρουσιάσουν τον Ιανουάριο στην επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. Ε, με αυτά και με αυτά, ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Βίβια Χόφμαν, αφού την καλημερίσω. Είναι Γενική Διευθύντρια τη DG ΕΑΚ e και θα μας παρουσιάσει αυτό το νομοθετικό πακέτο. Έχετε το λόγο για περίπου τα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, χαίρομαι που θα έχουμε αυτή την αλλαγή απόψεων. Ε, θα έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για τις καινοτομίες, ε, τα καινούργια στοιχεία ε, που επιφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση για την περίοδο 2021-2027 για το EIT. Το EIT δημιουργήθηκε ε, για να οθήσει τις δυνατότητες καινοτομίας, να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην καινοτομία και να αντιμετωπιστούν με πιο, μέσω μιας πιο συστηματικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε αυτά τα εμπόδια σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το EIT δημιουργήθηκε για να ξεπεραστούν κυρίως τα εμπόδια τα οποία παρεμποδίζουν την συνεργασία μεταξύ της, ε, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, ε, το ακαδημαϊκό. Έτσι λοιπόν αυτή η έννοια του να προωθηθεί ε, μια ευρωπαϊκή ένας ευρωπαϊκός χώρος γνώσης είναι στην καρδιά αυτής της προσπάθειας. Όπως ξέρετε το EIT εδώ και 10 χρόνια υπάρχει από το 2008 και η αποστολή του είναι να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την καινοτομία δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των, των ε, οικοσυστημάτων καινοτομίας τα μοντέλα του ε, δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια διότι ήταν πάντα επίκαιρα ε, δεν είναι δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογία. Αφορά όλη την αλυσίδα καινοτομία από την εκπαίδευση έω την αγορά. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι καινοτόμοι, επιχειρηματίε, οι φοιτητέ, ε, στα πλαίσια μιας προοπτική διαβίου μάθηση. Ε, στο μέλλον θα ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με την ανάγκη ενίσχυση τη δυνατότητα καινοτομία ε, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις κοινότητε καινοτομία που είναι συμπράξει ευρωπαϊκές ε, που όπου συμμετέχουν από 15 έως και 400 ε, εταίροι δίνονται υποτροφίες, τα kicks αυτά όπως τα λέμε ε, παρακολουθούμε τις εργασίες τους και βεβαίως διαδίδουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποτελέσματά τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τα βασικά στοιχεία της πρότασής μας, δηλαδή το EIT στα πλαίσια του οριζόντα 2021-2027, πάντα βέβαια με βάση τη δική του νομική βάση, θα ήθελα αρχικά να πω ότι η αρχή ε, που διέπει την πρότασή μας είναι ότι το μοντέλο πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, να κεφαλοποιήσουμε ε, τα δυνατά του σημεία και να βελτιώσουμε όπου χρειάζονται βελτι... βελτιώσεις. Έχουμε, προσ... Έχουμε προτείνει 3 δισεκατομμύρια για το σύνολο του EIT, ε αύξηση του προπολογισμού. Ποια είναι, ποια είναι η βασική τομή παρέμβαση. Τέσσερι τομεί κυρίω. Πρώτα απ' όλα, περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης σχετικών οικοσυστημάτων ανά την Ευρώπη. Δεύτερον, ενίσχυση της ε, των, των δεξιοτήτων καινοτομία και επιχειρηματικότητα στα πλαίσια τη διαβιωμάτιση, αυξάνοντα και τη δυνα... δυνατότητα των ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη να βρούμε νέε λύσει τρίτων ε, νέες, νέα αγαθά και υπηρεσίε για να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσει και τέταρτον να αναπτύξουμε συνέργειε και προσθέμενη αξία στα πλαίσια του ορίζοντα ε, τη Ευρώπη και άλλων ε, σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι συμπράξει ΚΙΚΣ ε, είναι συμπράξει και θα αποτελέσουν μέρο των ευρύτερων συμπράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, ακολουθήσουν λοιπόν τι βασικέ αρχέ και το, το κύκλο ζωή, τα σχετικά κριτήρια των συμπράξεων του Horizon έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια πιο ανοιχτή προσέγγιση όπως συμβαίνει και στα άλλα προγράμματα. Υπάρχει βεβαίως ευελιξία σε ό,τι αφορά το, μοντέλο KICS μέσω του κανονισμού EIT όπως ε, το προτείνουμε με μια σειρά από παρεκκλήσεις. Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το EIT. Πολύ σύντομα να τα συνοψίσω. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ανάγκη να είμαστε πιο συμπεριληπτικοί. Τα συστήματα καινοτομία να είναι πιο συμπεριληπτικά στην Ευρώπη και να είναι πιο βαθιά ριζωμένα στα τοπικά οικοσυστήματα. Αυτά τα τοπικά περιφερειακά συστήματα πρέπει οπωσδήποτε να έρχονται πιο κοντά στην καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε, όπω είπα επίση, τι δυνατότητε καινοτομία των αναδοτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φτάνουμε τώρα στον κανονισμό. Εμείς προτείνουμε μια αναδιατύπωση για τους εξής λόγους. Ο κανονισμός EIT εγκρίθηκε το 2008, ψηφίστηκε το 2008 και ο κανονισμός ανέφερε τα καθήκοντα, την αποστολή του EIT και το πλαίσιο λειτουργίας του. Το 2013 έγινε μια τροποποίηση για να ε, το ευθυγραμμίσουμε με την ορίζοντα 2020. Τώρα η προτινόμενη ε, αναθεώρηση γίνεται μέσω διατύπωση, έτσι ώστε να έχουμε πλέον μία νομοθετική πράξη με όλη την πρόταση, την αρχική πρόταση δηλαδή του 2008, την τροποποίηση του 2013 αλλά και την παρούσα πρόταση έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα των προτινόμενων αλλαγών. Επίσης προτείνουμε ο κανονισμός ε, να βασίζεται σε αρχές, να είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά τον χρόνο, δηλαδή να μην υπάρξει ανάγκη επιμέρους ε, τροπολογιών στο τέλος της κάθε περίοδου του πολιτικού νοσημικού πλαισίου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ευθυγράμμιση με τους στόχους του, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία και να ενισχύσουμε βέβαια τη συνέργεια με όλα τα άλλα σχετικά προγράμματα. Εμείς θεωρούμε ότι εφαρμόζοντας την αρχή της ουδετερότητας της χρονικής θα έχουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και σταθερότητα του κανονισμού EIT. Σε ό,τι αφορά τώρα τον, τη νέα ατζέντα για τη στρατηγική καινοτομία με βάση τον κανονισμό EIT, αυτή η νέα ατζέντα καινοτομίας ε, θα εγκρίνεται για κάθε επταετή ε, οικονομική περίοδο. Η παρούσα ατζέντα καλύπτει την παρούσα περίοδο έως δηλαδή το τέλος του επόμενου έτους γίνεται αναφορά στις μακροπρόθεσμες ε, ε, προτεραιότητες για το EIT και βεβαίως ε, βλέπουμε και τις δραστηριότητες στον τομέα σαν της εκπαίδευσης, πώς κατανέμεται ο προπολογισμός, η τιμή προτεραιότητας, ο χρονικός ορίζοντας για την επιλογή των διαφόρων προγραμμάτων. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στον κανονισμό. Πρώτα απ' όλα, πιο ανοιχτά πιο διαφανή KICS, το σύστημα χρηματοδότησης επίσης, το οποίο έχουμε ε, μεταρρυθμίσει έτσι ώστε να υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα, να επιτευχθεί πραγματικά μετά την 15η χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και βεβαίω υπάρχει και η σχέση μεταξύ του EIT και των KICS μετά από αυτή την περίοδο των 15 ετών. Τρίτον, η περιφερειακή διάσταση την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ενίσχυση των δυνατότητων και δυνατότητων καινοτομία των ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιλογή νέων ΚΙΚΣ και ιδιαίτερα δημιουργία ενός νέου ΚΙΚ για την ε, πολιτιστική βιομηχανία θα υπάρξει σχετικό διαγωνισμό για το 2021 και τέλος διακυβέρνηση. Εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε ε, το στρατηγικό ρόλο των ΚΙΚΣ διατηρώντας όμως το μοντέλο διακυβέρνησης και την εξαρτησία που τα τα διέπει ε, σε ό,τι αφορά τον τομέα του πολιτισμού και της ε, δημιουργίας γενικά. Εκεί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Ε. Οι κλάδοι αυτοί συνήθως είναι πολύ στενά συνδεμένοι με τα τοπικά οικοσυστήματα, όμως είναι κατακαιρματισμένος ο κλάδος αυτός και δεν υπάρχει επαρκής καινοτομία, δεν υπάρχουν δεξιότητες επιχειρηματικότητας επίσης. Αυτό είναι κάτι που θα έρθει να συμπληρώσει τα υπάρχοντα κήξη, Η δυνατότητα καινοτομία τη ανώτατη εκπαίδευση τώρα. Ε, αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένου τομεί παρέμβαση για το EIT, για την καινοτομία ε, και την επιχειρηματικότητα σε μια προοπτική διαβίου μάθηση, αυξάνοντα τι δυνατότητε των, των ε, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανά την Ευρώπη. Αυτό προτείνουμε. Γνωρίζουμε ότι ο αντίκτυπος της, της εκπαίδευσης ε, και των εργασιών του ΑΕΤ στον τομέα αυτών ενώνοντα ε, ε, τις, του τριγώνου έχουν περιθώριο βελτίωσης. Ε, επίσης γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο, το Συμβούλιο Ταγωνιστικότητας στις 29 Νοεμβρίου ενέκρινε μια γενική μερική προσέγγιση για τον κανονισμό EIT και μια έκθεση πρόοδου για το SIA και βεβαίως αναμένουμε τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Äh, Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Χόφμαν. Να περάσουμε τώρα στην συζήτηση με τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, και βεβαίως όλα τα μέλη που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις ή να συνεισφέρουν. Ο κύριος Έλερ πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί θα χρειαστεί να φύγω ε, νωρίς πρέπει να πάω στην Ήτρε. Πώς, ε, ποιο είναι η ουσία, το ζουμί του πράγματος. Πρώτη φορά βλέπουμε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής ε, Ήτρε και της Επιτροπής Πολιτισμού και λειτουργεί αυτή η συνεργασία. Ε, μέχρι τώρα δεν γινόταν λόγο ούτε για τα ΚΙΚΣ και δεν ήταν προτεραιότητα ούτε από την Κομισιόν ούτε από τα κράτη-μέλη. Επομένω, ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα έτσι ώστε να διατηρήσουμε αυτήν την, ε, αυτό το ενδεχόμενο, αυτή τη δυνατότητα ρεαλιστική. υπάρχουν θεσμικοί λόγοι που μπορεί να ζητήσουμε αναθεώρηση, αλλά στα με, εν, μέσω διαπραγματεύσεων ΠΔΠ ε, ξε, ξαναξεκίνησε η διαδικασία ή μπορεί να ξαναξεκινήσει η μπορει να επανέλθει ας πούμε η διαδικασια στην Κομισιόν ε, και ε, και μπορεί να επανέλθει ας πούμε στο κοινοβούλιο κάποια στιγμή στο δεύτερο μισό της θητείας αυτό που σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή οι υπουργοί δεν συμφωνήσουν να χρηματοδοτήσουν το ΑΕΤ με οποιοδήποτε ποσό, ε, τότε ε, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό όμως ε, που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να, να, έχουμε τις σωστές συζητήσεις για τον προπολισμό με το Συμβούλιο. υπάρχουν πολλοί θεσμικοί λόγοι για να ζητήσουμε αναθεώρηση, αλλά νομίζω ότι από πολιτική άποψη δεν έχει έννοια ε, ούτως ε, ή άλλως το Συμβούλιο δεν αποτελείται από ε, υπουργούς πολιτισμού αλλά από υπουργούς έρευνας. Επομένως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ε, για να υποστηρίξουμε ότι ε, αν πρέπει να κρατήσουμε ένα κικ ε, θα είναι αυτό για την βιομηχανία της δημιουργίας. Και δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε στο ε, προϋπολογισμό της Κομισιόν, αλλά στον δικό μας προϋπολογισμό. Βλέπετε ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου ε, αναφέρεται σε 1,8% επιπλέον, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει, αν δηλαδή συγκρίνεται με τα στοιχεία της πρότασης της Κομισιόν του 2018, θα έχουμε περίπου 120-150 εκατομμύρια ε, επιπλέον έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το ΚΙΚ. Άρα ε, ε, εάν δεχτούμε τα ποσά της Κομισιόν θα έχουμε πρόβλημα οικονομικό όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΚΙΚ. Επίσης, να είμαστε ρεαλιστές ξαναλέω. Εντάξει, υπάρχει μία έμφαση στην εκπαίδευση αλλά αυτό είναι προβληματικό σε σχέση με τις ε, ε, στη, σε σχέση με τις συνθήκες. Οι Υπουργοί Έρευνας ε, δεν τους αρέσει πάρα πολύ το EIT γιατί ε, υπάρχει πρόβλημα ή κάποιο πρόβλημα με τις συνθήκες. Ε, άρα, ναι, να λέμε ότι η εκπαίδευση παίζει ρόλο στο ΑΕΤ, αλλά ε, οι συνθήκες μπορούν να δώσουν πάτημα στο Συμβούλιο έτσι ώστε να μην προχωρήσει. Τρίτον, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα στοιχεία τα αριθμητικά, Εάν πάρουμε την πρόταση του Συμβουλίου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, ε, που δίνει κάποιο προϋπολογισμό που σταδιακά αυξάνεται, αυτό δεν λειτουργεί με το καινούριο ΚΙΚ. Αυτό που θέλουμε είναι εμπροστογενία κατά κάποιο τρόπο αύξηση, που μετά σταδιακά μπορεί να μειώνεται. Δηλαδή ένα προϋπολογισμό που δεν θα αυξάνεται σιγά σιγά, τότε γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουν αποτέλεσμα τα κίξε. Τα κίξε για να λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια στην αρχή. Εάν δηλαδή τα 50-60 εκατομμύρια που χρειάζεσαι τα δει στο τέλος, τότε δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί κανονικά το ΚΙΚ. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα τελικού ποσού. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι ο προϋπολογισμός να ξεκινήσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και μετά ενδεχομένως να μειώνεται σταδιακά. Γιατί αν δεν έχουμε ε, τον πρώτο χρόνο ε, τα κονδύλια στη διάθεσή μας για να δημιουργήσουμε ένα δημιουργικό κικ, δεν θα λειτουργήσει καλά. Ο ε, είμαι εισηγητής στην Ήτρα και για την πρόταση Horizon ε, και επομένως ε, πραγματικά εγώ επαγρυπνώ κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά τα συμφέροντα της Επιτροπής Πολιτισμού βεβαίως μπορώ να καταλάβω την έννοια της αναδιατύπωσης αλλά πραγματικά το ξαναλέω, εάν έχουμε αναδιατύπωση και αν ε, η Κομισιόν ε, χρησιμοποιήσει ακόμα μισό χρόνο, ας πούμε, ε, έτσι ώστε να ξαναδεί το κείμενο, τότε δεν θα προλάβουμε. Και αν δείτε και τα στοιχεία της ανακοινώσεις της ε, Φιλανδικής Προεδρίας μπορεί να υπάρχει ε, μία περικοπή του Horizon κατά 2,5 δις ε, και οπωσδήποτε αυτό θα είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Γι' αυτό ζητάμε να υπάρξει συνασπισμός δυνάμεων έτσι ώστε να ξεπεράσουμε ε, τον, ε, την πρόκληση, ε, τη θεσμική πρόκληση και να πω λοιπόν ότι δεν είναι πάρα πολύ λογικό να ζητήσουμε αναδιατύπωση γιατί θα, θα μας σφαγιάσουν στη συζήτηση για το πει Ευχαριστούμε Κρίστιαν Έλλερ. Ελπίζω να έχει αρκετό χρόνο και η κυρία Μπάντινγκ, γιατί επεκταθήκατε λίγο για να τοποθετηθεί εκείνη όπως πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ ε, τους παλιούς συναδέλφους ε, που με ενημέρωσαν. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτο σχετικά με την εκπαίδευση. Ενδιαφέρον θα ήταν αν μπορούσατε να μας ε, λέγατε τον, κάποια περισσότερα πράγματα σχετικά με τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης διαδικασίας ΚΙΚ, κυρίως όσον αφορά την, το θεματολόγιο της καινοτομίας. Ε, γιατί αυτό είναι το θέμα που με απασχολεί. Ε, υπάρχει... Υπάρχει η γραμμή 450, μάλλον ε, υπάρχουν τα 450 εκατομμύρια τα οποία λένε, αναφέρεται ότι θα προκύψουν από νέε δράσεις. τι σημαίνει αυτό ακριβώς, γιατί ε, μου εκφράστηκαν προβληματισμοί ότι ε, θα γίνει μια προσπάθεια παρέμβασης ε, στα συστήματα εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω, λαμβάνοντα υπόψη την αύξηση του προπολογισμού. Μ' αρέσει βεβαίω η ιδέα της τη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Φυσικά μας ενδιαφέρει και το θέλουμε αλλά το ποσό που αναφέρεται ίσως είναι υπερβολικά ε, φιλόδοξο. Αυτό που θέλω να μάθω είναι τι ακριβώς σχεδιάζεται για τα κράτη-μέλη και τι ακριβώς θα αλλάξει. Ε, όσον αφορά το ΚΙΚ για τη δημιουργική βιομηχανία και τον πολιτισμό, εξαιρετική ιδέα. Βεβαίως μπορώ να προτείνω ε, κάποιες τροποποιήσεις όσον αφορά ε, το, την διατύπωση θα πρέπει λίγο να τροποποιήσουμε την διατύπωση, ωστόσο είναι εξαιρετικά επικοδομητική ως ιδέα. Οι δημιουργικές βιομηχανίες, ας πούμε, ε, στην ε, ε, Αγγλία φέρνουν 10 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από ό,τι άλλες δραστηριότητες και επομένως μας ενδιαφέρει να είναι επιτυχημένη η διαδικασία αυτή σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, από τη στιγμή που προτείνονται δύο κίξ ταυτόχρονα, με διαφορά ε, τριών ετών, πιστεύετε ότι είναι, μπορεί να είναι βιώσιμα. Από τα κίξ που είχαν αυτόν τον ε, κύκλο των 14 ετών, μόναχα ένα ε, ήταν πραγματικά επιτυχημένο. Τα άλλα μπορεί να είχαν κάποιες επιτυχίες και για το κλίμα και για το, τα ψηφιακά, κάνουν καλή δουλειά, αλλά οικονομικά δεν είναι βιώσιμα. Έχουν μηδενικά εισοδήματα, δεν έχουν προκύψει από αυτά επενδύσεις. Ε, και επομένως αυτό το KXCI για το 22 και άλλο ένα το 25 ίσως δεν είναι βιώσιμα. Ε, μήπως θα ήταν καλύτερα το δεύτερο νέο KIC να το μετατοπίσουμε χρονικά λίγο αργότερα. Τέλος. Κοιτάξτε, ε, μια και έρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει πάντα ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Το κικ του κλίματος έχει Key National Center στο Λονδίνο. Αναφέρεται ότι το IT ενδεχομένως θα ξεπεράσει και τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό είναι κατανοητό, αλλά τι γίνεται ε, με τις, ε, με τις ε, τα εμπλεκόμενα ιδρύματα, τι θα γίνει σε περίπτωση Brexit. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Μελμπάρντα. Η ιδέα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι εξαιρετικά ε, καλή. Η ανάπτυξη της γνώση, τη ε, της καινοτομίας, των σχετικών κοινοτήτων που φέρνουν κοντά ε, τεχνολογικά ιδρύματα έρευνας, ακαδημαϊκό κόσμο, ε, επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργία νέων ε, προϊόντων, νέες αγορές, startup, όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα επιμέρους ε, κράτη-μέλη μπορούν να πετύχουν καλύτερα εάν ευρύτερα οι ευρύτερες περιοχές τους είναι ανταγωνιστικές. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε στην, στον ανταγωνισμό μεταξύ χωρών πρέπει να επενδύσουμε σε συμπράξεις μεταξύ χωρών. Η δυνατότητα καινοτομίας ε, και κεφαλοποίησης ε, των καινοτομιών αυτών ε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δυνητικό, είναι απαραίτητο να συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν, να συνεχιστεί το έργο του EIT. Γενικά υποστηρίζω την κατεύθυνση που ακολουθείτε. Πιστεύω ότι το πακέτο αναθεώρησης για το, το για, την, ε, για το EIT ε έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Εγώ εκπροσωπώ τον τομέα του πολιτισμού και καλωσορίζω το γεγονό ότι η ατζέντα για τη στρατηγική καινοτομία αναφέρεται στον τομέα τη δημιουργία και του πολιτισμού ω ε, τομεί προτεραιότητα για, νέα, για νέε συμπράξει με έναν διαγωνισμό που θα ξεκινήσει το 2021. Βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και μια αντίσταση ε, από μια σειρά από κράτη μέλη στο Συμβούλιο που δεν επιθυμούν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίξ και το να ξεκινήσει σε δύο χρόνια. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου για τη γεωγραφική ισορροπία. Εγώ προέρχομαι από μια σχετικά μικρή χώρα της ε, Κεντροανατολικής Ευρώπης ε, τα κέντρα αυτά βρίσκονται κυρίως ε, ε στις πρώην παλαιές χώρες, στα 15 πρώτα κράτη-μέλη, αν δούμε και την, τον χώρα, τη χώρα των επιλέξιμων κρατών μελών, ε, αν δούμε και τα scoreboard, θα πρέπει να γίνει πιο ευρύς ο κατάλογος επιλεξιμότητας, δεν περιλαμβάνονται μόνο ε, τα μικρά κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 40% των ε, εργαζομένων προέρχονται από αυτές τις επιλέξιμες χώρες ε, σε ένα, στα πλαίσια ενός τέλειου ας πούμε σενάριου θα μπορούσε κανείς να ζητήσει μεγαλύτερο προπολογισμό για το Ινστιτούτο. Βεβαίως υπάρχει και η πολιτική πραγματικότητα Ήδη μια μικρή αύξηση λοιπόν θα ήταν επιτυχία. Επιπλέον πιστεύω πρέπει να περιοριστεί ο λίστο, η λίστα επιλεξιμότητας και να βασιστούμε στον, ε, αντίστοιχη λίστα του Horizon. Πάντως ε, με εμπνέει το έργο του Ινστιτούτου αυτού και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη για το μέλλον. Ως και ως εισηγήτρια αναμένω να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν έρθει και άλλοι και ο βλέπω. Δεν ξέρω αν θέλετε το λόγο ή αν θέλετε να περιμένετε ε, την παρέμβαση του επόμενου μιλητή. Ο κύριος Ρουίθ Ντεβέσα έχει το λόγο. Ναι, ήθελα να τελειώσει ο γύρος ε, για να μην ε, παρενοχλήσω. Κύριε Γεωργούλη, όχι, ωραία. Ε, κυρία Γένμπο, ε, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη, τι είδους ε, εταίρους ε, ζητάτε από τη βιομηχανία. Δεύτερον, ε, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί ε, ΚΙΚ ε, για τις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας και τρίτον ποια θα είναι η θέση και της πρωτοβουλίας στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στα πλαίσια του έρασμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρουίς Δεβέσα. Θέλετε τώρα να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Uh, <clears throat> we are, um, uh, συζητούμε το ε, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε και κάποια άλλα θέματα σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που έχουμε ε, συγκεκριμένα και για, την, για τον πολιτισμό ε, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα κομμάτι της ε, ε, παραγωγής, ας πούμε, που συμβάλλει πολύ στην ευρωπαϊκή οικονομία. I think, um, you know, um... We are of... Σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε αυτήν την προσέγγιση. Ε, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια καλή έκθεση και ευχαριστούμε την εισηγητή. Mr. Georgoulis, do you want to take the floor? Κύριε Γεωργούλη, θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Ε, πολύ ωραία. Sorry, Mrs. Ward. Julie. Uh, okay, thank you very much. Κυρία Ward, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Και πραγματικά χαίρομαι που η δημιουργική βιομηχανία, ο κλάδος της δημιουργίας είναι κάτι που μας απασχολεί πλέον και αρχίζει να εμποτίζει και άλλες σφαίρες δραστηριότητας. Εγώ ήμουν ένθερμη υποστηρίκτρια του STEAM, ατμός αντί για STEM, τα προηγούμενα αρχικά. Και θα ήταν καλό πραγματικά οι τέχνες και ο πολιτισμός να ξεπεράσουν τα στενά όρια στα οποία τους έχουμε τοποθετήσει και να επιστρέψουν εκεί που πρέπει. Μιλάμε για καινοτομία, για επιχειρηματικότητα και ήθελα απλώς να μου πείτε αν η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει διότι το επιχειρήν αυτό καθεθώ είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Όμως το κοινωνικό επιχειρήν, η κοινωνική επιχειρηματικότητα ακόμα δεν ε, γίνεται κατανοητή από τον κόσμο. Νομίζουν ότι είναι φιλανθρωπία. Εγώ είμαι υπεύθυνη μιας κοινωνικής επιχείρησης και είναι κανονική εταιρεία ε, πρέπει να λειτουργήσει και να είναι βιώσιμη βάσει επιχειρηματικών μοντέλων, των business model που λέμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να το συζητήσει λοιπόν αυτό και να το λάβει υπόψη. Έχουμε τώρα μια πολύ καλή ευκαιρία για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ε, να το δούμε ως ε, μοντέλο για εταιρεία, για επιχείρηση, για κόσμο που, είναι πολύ, που απασχολείται στον τομέα της δημιουργίας. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ ήθελα να σχολιάσω κάποια σημεία. Ιδίω το κεκ για, για την ε, βιομηχανία της δημιουργίας. Είναι σαφές ότι ο τομέας της δημιουργίας ε, είναι υπεύθυνο για το 40% του ΑΕΠ στην Ευρώπη και για πολλές θέσεις εργασίας. Είναι υπεύθυνο για πολλές, δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης και πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι νέες τεχνολογίες. Είναι πολλά τα στοιχεία που χάρη στον κλάδο της δημιουργίας επηρεάζονται και δίνουν μια όθηση ή παίρνουν μια όθηση μέσα από την ε, δημιουργική βιομηχανία. Όπως και ο κινηματογράφος και άλλοι τομείς, η μουσική, έχουν παίξει ζωτικό ρόλο με τη χρήση νέων τεχνολογιών και αυτό βοηθάει να παραμείνουν στην εμπροστοφυλακή. Έτσι θεωρώ ότι είναι ε, εντελώς σημαντικά τα στοιχεία του Ινστιτούτου της Τεχνολογίας και θα πρέπει πραγματικά να δοθεί μια ε, ισχυρότερη όθηση με την κατάλληλη χρηματοδότηση, την κατάλληλη πρικοδότηση. Πρέπει ένα κικ ε, κατάλληλο να προβλεφθεί ως κονδύλι στη χρηματοδότηση και να μπορέσουν και τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη την ε, δράση του Ινστιτούτου. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου Διότι ακριβώ στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα τη ε, Δημιουργική Ευρώπη, το Creative Europe, του Horizon 2020 και σε ό,τι αφορά την πληροφορική και την τεχνολογία, μαζί με το δεδομένο ότι πρόκειται να γίνει το Brexit, πρέπει να φροντίσουμε παρόλα αυτά τα στοιχεία να λάβουν τα απαραίτητα κονδύλια μέσα από τον προπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, ως μέλη της Επιτροπής και ασχέτως πολιτικής ομάδας να ζητήσουν ακριβώς ένα τέτοιο ισχυρό για την δημιουργία τη μηχανία στην Ευρώπη. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος τον ε, λόγο για το θέμα αυτό. Οπότε να δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Χόφμαν για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα επικοδημητικά σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, υποστήριξη και για, το δημιουργικά, ε, για τα δημιουργικά κίκ. Ε, πραγματικά, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, αυτοί, αυτές οι, αυτοί οι κλάδοι ε, έχουν πραγματικά πολύ μεγάλες ικανότητες. Από την άλλη πλευρά όμως και παρά τις πολλές δυνατότητες εξακολουθούν να υπάρχουν προσκόμματα και φρακτήρες φραγή. Ε, θεωρούμε ότι τα CCIs δεν έχουν ακόμα ε, εγγραφεί στα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι πρέπει όντως να υποστηριχθούν ε, μέσω αυτών των καινοτόμων συστημάτων και μέσω συμπράξεων με άλλους δυναμικούς εταίρους. Όσον αφορά την εκπαίδευση, πιστεύουμε ότι, ότι ο, οι, οι πλευρές όλες του τριγώνου πρέπει να είναι ε, δυνατές έτσι ώστε το ίδιο το τρίγωνο στο σύνολό του ε, να είναι ε, δυνατό. Δεν προτιθέμεθα εμείς βεβαίως να παρέμβουμε ε, στην οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών. Ωστόσο, αυτό που θέλουμε ε, είναι ε, ένα εργαλείο το οποίο σε ολόκληρη την Ευρώπη θα παρασχεθεί στην τριτοβαθμία εκπαίδευση, πράγμα που σημαίνει ότι και στην ανώτερη εκπαίδευση θα βρεθούν και νέοι εταίροι και νέες συμπράξεις. Αυτός είναι ένας στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, Πιστεύουμε ότι ένα ικανό κομμάτι του προϋπολογισμού θα πρέπει να δοθεί. Δεν θέλω όμως να μιλήσω εν για τον προϋπολογισμό τώρα. γιατί ε, ε, αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση. Οπωσδήποτε εγώ θα μεταφέρω όλα τα ε, στοιχεία που άκουσα εδώ. Όταν Όταν θα έχει εγκριθεί και η έκθεση του Κοινοβουλίου, τότε ε, θα μπει σε λεπτομέρειες ε, και η Κομισιόνα. Όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα, κατά τη δική μας άποψη, αυτή είναι μια σημαντική αρχή. Ε, υπήρχε από την αρχή ε, η αρχή αυτή στον, στο κείμενο, τώρα όμως την ενισχύουμε. Ε, η κεντρική ιδέα δεν είναι διαρκώς να χρηματοδοτούμε τα κίξε, αλλά κάποια στιγμή να βρουν τα κίξε άλλους ε, τρόπους και πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, δεν θέλουμε τα κίξε να είναι απολύτως αποσυνδεδεμένα από άλλες ε, πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την περίοδο των 15 ετών. Γι' αυτό ε, ε, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν δεσμοί και μάλιστα δίνουμε την δυνατότητα ακόμα και μετά τη 15 ετη περίοδο τα ΚΙΚΣ να μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες. Όσον αφορά τώρα τους, τα νέα ΚΙΚΣ, ο προϋπολογισμός παραμένει ίδιος εάν είμαστε πολύ φιλόδοξοι όσον αφορά τη δημιουργία νέων κίξ και λέμε ότι ένα δεύτερο ε, θα ε, πρέπει να ε, προταθεί στην, εντός της περίοδου πι τότε θα πρέπει οπωσδήποτε τα πρώτα τα πρώτης γενεάς ΚΙΚΣ ε, μέχρι το 2024 να ε, αποδείξουν ότι έχουν ε, οικονομική βιωσιμότητα. Για, τον, για τη χρηματοδότηση των ΚΙΚΣ έχει προβλεφθεί μία μειούμενη συμβολή έτσι ώστε ακριβώς να τους δώσουμε τα κίνητρα στα κίξ αυτά για να δραστηριοποιηθούν. Αυτή είναι η έννοια. Όσον αφορά την περιφερειακή διάσταση, πράγμα πολύ σημαντικό, συμφωνούμε απολύτως ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε η γεωγραφική προσέγγιση να ε, διευρυνθεί. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει το, το, να γίνει υποχρεωτικό. Είναι αυτά τα Regional Innovation Scheme. Θέλουμε να γίνει υποχρεωτικό ε, εντός των πλαισίων της μακροχρόνιας στρατηγικής των ΚΙΚΣ ε, και προτείνουμε ότι τουλάχιστον 250 εκατομμύρια να ε, δοθούν στις δραστηριότητες ΡΙΣ πέρα από το 20% το οποίο ε, δίνεται στην εκπαίδευση και που ε, αφορά την ε, μετάβαση στην καινοτομία. Include the cases that uh, it should be a variety, um, bigger company. βεβαίως θέλουμε εταιρείε, μικρομεσαίες εταιρείες από διάφορους τομείς Όσον αφορά τώρα την ε, σχέση με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, η κοινότητα IT έχει ήδη αναπτύξει τεχνογνωσία σε τομείς που σχετίζονται και με τα ε, πανεπιστήμια, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως ας πούμε και ένα τόμα παιδαγωγική και άλλα και πιστεύουμε ότι πραγματικά πρόκειται για μια διαδικασία το συμπληρωματική προς τα πανεπιστήμια. Όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, έχω να πω τα εξής. Γίνεται αναφορά στην ε, κοινωνική καινοτομία ε, στα πλαίσια των ΚΙΚ και της, ε, του κλάδου της δημιουργικής παραγωγής. 2-3, 2 τρίτα των, ε, των Κίξε ε, ε, θα είναι επιλέξιμα. Βεβαίως, εάν δεν υπάρξει συμφωνία... UK... Um, θα χρηματοδοτηθεί από τα, σε περίπτωση του Brexit θα προκύψει χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη ε, αλλά ε, ε, θα εξακολουθήσουν ε, τα πανεπιστήμια να είναι επιλέξιμα για την χρηματοδότηση και θα πρέπει παρόλα αυτά να διατηρηθεί αυτό το ποσοστό των δύο τρίτων που θα προέρχεται από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια στα ΚΙΚΣ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ολοκληρώθηκε η ανοιχτή συνεδρίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Χόφμαν για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι δεν έχουν άδεια να παραμείνουν στην αίθουσα να την εγκαταλείψουν ησύχως για να ξεκινήσει η συνεδρία κλεισμένο των θυρών. Also bitte alle die, die nicht zum Parlament gehören. Όσοι δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εδώ στην αίθουσα, παρακαλώ να αποχωρήσουν για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Βουλευτέ, βοηθοί, όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην ε, συνεδρία των συντονιστών, παρακαλούμε να αποχωρήσουν.